ή εάν μέχρι την δημοσίευση των πρακτικών δεν έχουν υπάρξει αντιρρήσεις θεωρούνται πως εγκρίνονται. Η κυρία Αγγέλικα Βέρτμαν μου ανακοίνωσε πως ε, προσχώρησε στην ομάδα των φιλελευθέρων. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 κατέθεσε μια αιτιολογημένη γνώμη η οποία